ότι ο Μίλος Λαφράνστο, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 2016 σε ηλικία 62 ετών. Ο κ. Ράνστοφ ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2003 το 2016 ω μέλος της GUE-NGL. Ήταν αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Βιομηχανία, Έρευνα και ενέργεια και μέλος της αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest και την αντιπροσωπεία με την Ουκρανία. Ήταν δόκτωρ φιλοσοφίας ο Μίλος Φράνστοφ, ήταν γνωστός ε, συγγραφέας βιβλίων και μελετών και ήταν ιδιαίτερος ε, εμπειρογνώμος στα θέματα της μεταρρύθμισης για τον Μάξ και για τα θέματα της αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας. Σας παρακαλώ να κρατήσετε ενός λεπτού στη γη για τον απολεσθέντα συνάδελφό μας.